Ε, μου ε, ε, κατέθεσε την παρέτησή του από τις 15 Μαρτίου, διαπιστώνει το Κοινοβούλιο τη χειρία της έδρας και ενημερώνει τις αρμόδιες εθνικές αρχές. Οι αρμόδιες ισπανικές αρχές με ενημέρωσαν ότι εκλέγεται ο κύριος Μιγγέλ Ουρμπάν Κρέσκο από την 5η Μαρτίου 2015 και αντικαθιστά συνάδελφο την κυρία Τερέζα Ροντρίγκε Ρουμπίου. Το Κοινοβούλιο ε, σημειώνει αυτή την ανακοίνωση. Καλά, ε, σορίζω το συνάδελφο και του ανακοινώνω ότι συμμετέχει πλήρω στι συνεδριάσει Ολομέλεια και των οργάνων του Κοινοβουλίου με την επιφύλαξη των σχετικών άρθρων του κανονισμού. Στις 24 Φεβρουαρίου συνεδρίασε η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων και ήλεγξε σύμφωνα με τον κανονισμό